Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στην ε, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ρέντινγκ. Άρχεται η συνεδρίαση. Ως ε, πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη έχουμε το ενέκθεση του κυρίου Σαλαβράκου, της δραστηριότητας του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2012. Για άλλη μια φορά, μετά από την επίσημη έναρξη της ε, συνεδρίασης, Καλωσορίζω τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον κύριο ε, Διαμαντούρο. Καλώς ήρθατε. Και... Έχετε κάποιο σημείο διαδικαστικό? Κύριε Πρόεδρε, Καταρχάς, καλωσορίσατε, πολλές ευχές. Νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας να καλωσορίσουμε τον διαπραγματευτή Κατόπιν πρωτοβουλίας της Ολυγιακής Επιτροπής ε, Γιορτάζουμε στην Ιταλία για να θυμηθούμε το ρεκόρ στο Μεξικό του Πιέτρου, το, ρεκόρ του Πιέτρου Βενέα. Το ρεκόρ αυτό διήρκεσε 17 χρόνια και το κατέριψε μόνο ο Μάικλ Τζόνσον. Ο Μενέα πέθανε τον προηγούμενο Μάρτιο σε ηλικία 60 ετών. Θα ήθελα λοιπόν να θυμίσω το Μενέα γιατί από το 89 μέχρι το 2004 υπήρξε μέρος του Κοινοβουλίου. Συνέγραψε, συνέταξε την έκθεση για τον αθλητισμό και έδωσε ολόκληρο αγώνα κατά του ντόπινγκ πιστεύοντας σε καθαρό αθλητισμό ελεύθερο από τους οργανισμούς εκείνους που δεν προάγουν το σωστό πνεύμα του αθλητισμού. Η νίκη του Μενέα το 79 αποτέλεσε πηγή μεγάλης χαράς και περηφάνειας για την Ιταλία. Η ε, δύναμη του Μενέα που κατάφερε να προπονηθεί στον δρόμο τον οδήγησε στο να την ε, κορυφή ενσαρκώνοντας τις, ε, τις, ε, τους αγώνες μιας ολόκληρης γενιάς. Σήμερα γίνονται πάρα πολλοί εορτασμοί στην Ιταλία για να θυμίσουν τον Μενέα. Θα γίνουν αγώνες με θεσινούς και σημερινούς αγωνιστές αλλά πιστεύω ότι εδώ σε αυτή την αίθουσα θα πρέπει να το βοηθήσουμε φόρο τιμής και να το θυμηθούμε γιατί υπήρξε ένας βουλευτής ο οποίος προήγαγε την ιδέα του αθλητισμού και νομίζω ότι είναι σκόπιμο να τον θυμηθεί αυτό το Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας, κύριε Σιλβέστρης. Φτάνουμε λοιπόν στο πρώτο σημείο της σημερινής διάταξης, ε, την έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το 2012. Για τέσσερα λεπτά ο κύριος Αλαβράκος έχει το λόγο ως ε, εισηγητής ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και χαίρομαι ιδιαίτερα που σας έχουμε πάλι κοντά μας. Εύχομαι να μην έχετε άλλο ατύχημα. Ε, αισθάνομαι την υποχρέωση να επενέσω τον διαμεσολογητή μας τον κύριο Διαμαντούρου ο οποίος έχει εκπροσωπήσει και υπηρετήσει επάξια το θεσμό τα τελευταία δέκα χρόνια ένα θεσμό ο οποίος ενώνει τους Ευρωπαίους πολίτες και τους δημιουργεί ένα ασφαλές αίσθημα καταφυγής θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδεις συγητές για τις τροπολογίες τους και για την επικοδομητική συνεργασία τους προς ολοκλήρωση της ετήσιας έκθεσης για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή του έτους 2012. Ως εισηγητής της έκθεσης σημειώνω την πρόοδο που έχει επιτελέσει ο θεσμός, διαπιστώνοντας ότι σε σχέση με πέρσι είναι ακόμη μεγαλύτερη. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να σας αναφέρω κάποια σημεία της εκθέσεως που αναδεικνύουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί συγκεκριμένα το 2012 χιλιάδες υπήρξε μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά καθώς ο αριθμός των ερευνών που διεξήχθησαν και περιόθησαν ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. οι συνολικές έρευνες που ξεκίνησαν σημείωσαν αύξηση κατά 18% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του. 2011. Ο αριθμός των ερευνών που περαιώθησαν αυξήθηκε κατά 23% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά όπως και το 2011, ο διαμεσολαβητής εξυπηρέτησε άμεσα περισσότερο από 22.000 πολίτες, εξετάζοντας τις αναφορές τους, απαντώντας στα αιτήματά τους και παρέχοντας συμβουλές μέσω του διαδραστικού οδηγού στον δικτυακό τόπο. Χάρη στις χρήσιμες συμβουλές που παρέχει ο οδηγός, ο αριθμός των αναφορών που ήταν εκτός της αρμοδιότητας του διαμεσολαβητή ήταν χαμηλότερος στις τελευταίες δεκαετίες 69% των ερευνών περατώνεται εντό ενό έτου, ποσοστό μάλιστα που είναι ελαφρά βελτιωμένο σε σχέση με το 2011 που είχαμε 66%. Οι περισσότερε έρευνε που ξεκίνησαν το 2012 αφορούσαν μορφέ εικαζόμενη κακοδιοίκηση σε ζητήματα νομιμότητος, πρόσβαση σε στοιχεία και πληροφορίε, ακριβοδίκαιε μεταχείρισης και τήρηση των ευλόγων προθεσμιών κατά την ύψη των αποφάσεων μεταξύ άλλων η αρμοδιότητα του διαμεσολαβητή για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αναγνωρίστηκε στην απόφαση του συμβουλίου η οποία επικύρωσε το σχετικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής ένωσης δυνάμει της σύμβασης των ηνωμένων εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. ο διαμεσολαβητής συνεργάζεται με τέσσερα άλλα όργανα μεταξύ των οποίων η επιτροπή αναφορών του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου με στόχο να προστατεύσει να προάγει και να παρακολουθήσει την υλοποίηση της σύμβασης. Κύριε συνάδελφοι συγχαίρω θερμά τη νέα διαμεσολαβητή την κυρία Ωρέλη, για την εκλογή της και επιθυμώ να της ευχηθώ το καλύτερο για τα νέα της καθήκοντες. είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει το όραμα του απερχομένου ευρωπαίου διαμεσολαβητή με αποφυσίωση με δυναμισμό και με απότερο στόχο το συμφέρον των ευρωπαίων πολιτών. εκφράζω στον ε, κύριο διαμαντούρο την ευγνωμοσύνη μου για το υποδειγματικό έργο ως ευρωπαίος διαμεσολαβητής το οποίο πραγματοποίησε την τελευταία δεκαετία και για τα αποτελέσματα που πέτυχε καθιστώντας την ευρωπαϊκή ένωση δικαιότερη και διαφανέστερη. σαν έλληνας είμαι υπερήφανος γι' αυτό. του εύχομαι να έχει καλή υγεία ατομική και οικογενειακή ευτυχία και επιτυχία στις μελλοντικές επιδιώξεις του. ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Διαμαντούρας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν να διατυπώσω τις παρατηρήσεις μου, θα ήθελα να σας καλωσορίσω Χαίρομαι ιδιαίτερα που χαίρεται άκρα υγείας. Αυτό με ικανοποιεί ιδιαίτερα. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, αυτή είναι μια στιγμή πολύ συγνητική για μένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρασουλιάσω την ετήσια έκθεσή μου για το 2012. Θα ήθελα να εκφράσω καταρχάς τις θερμότατες ευχαριστίες μου στον εισηγητή κύριο Σαλαβράκο για την τόσο ενδελεχή του έκθεση για τις δραστηριότητες του διαμεσολαβητή αλλά και την Επιτροπή η οποία πραγματικά υπήρξε μια πηγή έμπνευση για μένα κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον κύριο Σαραβράκο για τις παρατηρήσεις που διατύπωσε σε προσωπικό επίπεδο. Πραγματικά με άγγιξαν βαθιά. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, το 2012 22.000 ε, πολίτες βοηθήθηκαν από τον διαμεσολαβητή 19.000 έλαβαν ε, στοιχεία μέσω του διαδραστικού δικτύου. Βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους πολίτες να καθοδηγούνται από τον φορέα που χειρίζεται αυτές τις καταγγελίες και με αυτόν τον τρόπο να μην χρειάζεται να αναζητούν μόνοι τους το κατάλληλο φορέα. Το 12 έλαβα 2.242 καταγγελίες από πολίτες, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, οργανώσεις, ενώσεις και άλλους οι 465 έρευνες που ξεκίνησαν το 12 αντιπροσωπεύουν μία αύξηση κατά 18% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτός ακολουθεί μία αύξηση που παρατηρήθηκε κατά 18% το 11. Υπάρχει μία τάση που επιβεβαιώνεται από τη μείωση στον αριθμό των καταγγελιών που ελήφθησαν εκτός της θητείας. Το 2012 ο αριθμός αυτών των καταγγελιών ήταν 1720 ε, που είναι ο χαμηλότερος βαθμός σε διάστημα 10 ετών. Αποδίδω αυτή την ε, επιτυχία στον διαδραστικό οδηγό που ανέφερα πριν από λίγο. 290 καταγγελίες, 390 καταγγελίες έκλεισαν. Σε πολλές περιπτώσεις ε, υπήρξε συμφωνία για μια φιλική λύση ή έγινε δεκτή μια σύσταση. Περισσότερες από τις άλλες περιπτώσεις έκλεισαν ε, με τη διαπίστωση ότι δεν χρειάζονται περαιτέρω έρευνες. τα θεσμικά όργανα δέχτηκαν ένα σχέδιο σύσταση σε 9 από τι 56 περιπτώσεις ενώ οι άλλε 47 περιπτώσει έκλεισαν με παρατηρήσει Σε 30 περιπτώσει έκανα περαιτέρω παρατηρήσεις για να μπορέσω να βελτιώσω την όλη κατάσταση. Αξιότιμα μέλη, το 2012 για πρώτη φορά μπορέσαμε να δώσουμε μία απάντηση στο ερώτημα του πόσο καλά συνεργάζονται οι θεσμοί με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν τη δική τους απόδοση. Σε δύο δημοσιεύσεις ε, που έγιναν πέρσι ε, μια έκθεση συμμόρφωση και μια άλλη δημοσίευση, διαπιστώσαμε ότι το 82% των, 82% των περιπτώσεων οι θεσμοί συμμορφώθηκαν με τι υποδείξεις του διαμεσολαβητή. Ήθελα επίσης να πω ότι το ποσοστό συμμόρφωσης για την Επιτροπή ήταν ακριβώς το ίδιο επίπεδο 82, δηλαδή 100. Η διαφάλιση υψηλών επιπέδων συμπεριφορά στα θεσμικά όργανα αποτελεί κομβικό σημείο της αποστολής του διαμεσολαβητή. Το 2012 μετά από μία δημόσια διαβούλευση καθορίστηκαν ορισμένες αρχε Οι πέντε αρχές αποτελούν μία ευσύνοπτη δήλωση ε, τι αναμένουν οι πολίτε από τι δημόσιε υπηρεσίε. Καταρχά δέσμευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του πολίτε, δεύτερον κυριότητα, τρίτον αντικειμενικότητα, τέταρτον σεβασμό για του άλλου και πέμπτον διαφάνεια. Αυτέ οι αρχέ λαμβάνουν υπόψη τι βέλτιστες πρακτικέ στι χώρε μέλη και μεταξύ των άλλων θα πρέπει να βοηθήσουν του δημόσιου υπαλλήλου να καταλάβουν την πληθώρα των ε, ε κανονισμών που διέπουν τι του. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα ε, μέλη, επειδή θα συνταξιοδοτηθώ στο τέλος του μήνα, θα ήθελα να <clears throat> σας πω ε, ποιες ήταν, ποια ήταν τα επιτεύγματα του θεσμού στον οποίο με εκλέξατε τρεις φορές την προηγούμενη δεκαετία. Τα τελευταία δεκάμιση χρόνια ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής επελήφθη 33.000 περιπτώσεων και ξεκίνησε 3.500 ε, εντελεχείς Έρευνε σε περιπτώσει κακή διοίκησης. Κατά τη διάρκεια του ιδίου χρονικού διαστήματο, η διοίκηση έγινε περισσότερο φιλική προ το ε, πολίτη, περισσότερο στραμμένη προς τι υπηρεσίες και περισσότερο διαφανή. Είμαι πεπισμένο ότι η ανεξάρτητη ε, εργασία του διαμεσολαβητή συνέβαλε έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια διοικητική κουλτούρα. Επειδή είχαμε αυτά αποτελέσματα σε πολλού τομεί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, θέματα δεοντολογία, ας πούμε, σύγκρουση συμφερόντων και τα δικαιώματα των πολιτών. Από, την, από τότε που έδειξε εφαρμογή η συνθήκη τη Λισαβόνα και η χάρτα των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων έγινε δεσμευτική, ο διαμεσολαβική δραστηριοποίηση στον τομέα των δικαιωμάτων των πολιτών. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την πρωτο, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία, η υποχρέωση διεξαγωγή του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών και αυξημένη συμμετοχή των πολιτών συμπεριλαμβανομένων και των ε, δημοσίων διαβουλεύσεων. Ο μεσολαβητή πήρε μέρο με πολλού τρόπου στη λήψη αποφάσεων και στη διαμόρφωση ε, ε, απόψεων. Ε, ένα σημαντικό μέρος της εργασίας μου αφορούσε προσαρμογή έτσι ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη μεταρρύθμιση του καταστατικού με βάση την, ε, ε, την, δημιουργία του, της θέσης του διαμεσολαβικής στη Τουρκία, ε, τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ενίσχυση του δικτύου Ευρωπαίων Διαμεσολαβητών και την παροχή πληροφοριών και συστάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η προώθηση μιας διοικητικής κουλτούρας συνεπάγεται μια ηθική δέσμευση και από πλευρά του Κοινοβουλίου και των άλλων θεσμικών οργάνων. Ζητά από το ε, διαμεσολαβητή να κάνει επίδειξη φαντασίας εκ των προτέρων αντίδρασης και μια συγκεκριμένη αντίληψη σε ό,τι αφορά τα θεσμικά όργανα. Πάνω απ' όλα να προωθηθεί μια κουλτούρα συγκεκριμένη που συνεπάγεται δέσμευση και διοικητικές ικανότητες για να υιοθετηθούν στρατηγικές που συνδέονται με ε, υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Αυτό αποτελούν την βασική βάση όπου θα στηριχθεί το ηθικό και πολιτικό κεφάλαιο που είναι απαραίτητο για το διαμεσολαβητή για να σταθεί στο ύψος των προσδοκιών ε, των πολιτών ε, αφού θεωρείται ένα αντίβαρο στην εκτελεστική εξουσία να μπορεί ε, δηλαδή να έχει την ικανότητα ουσιοδός να συμβάλλει στην κατανόηση των νόμων και στη βελτίωση το χαρακτηριστικό της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι θα είχε λίγη πρόοδος δίχως τη συνεργασία του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Το, το προσωπικό ξεκίνησε έναν ε, δημιουργικό διάλογο και αυτό αποτέλεσε ένα σημαντικό στοιχείο της άποψής μου ότι η διαμεσολαβητής δεν θα πρέπει να θεωρείται ως μια θεσμική έκφραση μιας κουλτούρας ε, καταγγελιών ο στόχος ήταν να προωθηθεί μια κουλτούρα παροχής υπηρεσιών και σεβασμού των δικαιωμάτων των πολιτών. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επιτρόπους ε, που συνέβαλαν σε αυτό τον τομέα καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Τις περισσότερες περιπτώσεις ε, συνεργάστηκα μαζί μου στην προώθηση της ε, αρχής μιας κουλτούρας υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ε, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την παρουσία της κυρίας Ρέντινγκ για να υπογραμμίσω τον τρόπο με τον οποίο συνέβαλε και εκείνη και τον τρόπο με τον οποίο με υποστήριξε στο παρελθόν. Τέλος, θα ήθελα να αναγνωρίσω το βασικό ρόλο του Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα της Επιτροπής Αναφορών, και την υποστήριξή του προς τον θεσμό του διαμεσολαβητή. Το Κοινοβούλιο εξασφάλισε τους απαραίτητους πόρους για να μπορέσει να συνεργαστεί αποτελεσματικά και παρήχε ε, στήριξη στον διαμεσολαβητή για να μπορέσει να προασπίσει τα δικαιώματα των πολιτών. Υπήρξε μια κοινή προσπάθεια που πιστεύω ότι ε, ε, οδήγησε σε θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες. Θα ήθελα να κάνω ορισμένε σκέψει ό,τι αφορά τι προκλήσει για το μέλλον. Το Κοινοβούλιο, εν τη συλλογική του σοφία, εξέλεξε την κυρία Ορέιλι. Ε, η κυρία... Ρέιλι είναι προετοιμασμένα για όσα επίγενται. Νομίζω ότι διακρίθηκε και σε επίπεδο εθνικό και σε επίπεδο διεθνές. Προείδευσε ε, ε, ε, στο εσωτερικό της, ε, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη χώρα της, ενώ διεθνώς διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και της Ένωσης των, του Βρετανών και Ιρλανδών ε, διαμεσολαβητών. Τέλος, επειδή είναι η πρώτη γυναίκα διαμεσολαβητής, ε, χαρακτηρίζεται από την συναισθηματική ε, νοημοσύνη που χαρακτηρίζει το φίλο τη είναι απόλυτα προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει τι προκλήσει του ρόλου τη. Ένας από τους τις προκλήσεις αυτές, μία από τι προκλήσει αυτέ είναι η οικονομική στενότητα. Αυτό είναι κάτι που θα κληθεί να αντιμετωπίσει αρκετές φορές. Μία άλλη πρόκληση είναι η προσαρμογή στις τεχνολογικές αλλαγές, τα οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Το θέμα της γύρασης του πληθυσμού, καθώς και άλλα προβλήματα συμπεριλαμβανομένες και της μετανάστευσης αυτές οι προκλήσεις χαράσουν τη σχέση μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Οι πολίτες έχουν πάρα πολλές προσδοκίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξαρτώνται από δύο παραμέτρους. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα εργαλεία που, έχουμε, τα εργαλεία που έχουν για να τα κοινοποιήσουν όλα αυτά. Η πρόκληση για τον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή είναι το να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών και παράλληλα να έχει απόλυτη συνείδηση των πιέσεων και των περιορισμών. Θα ήθελα να ευχηθώ στον διάδοχό μου ό,τι καλύτερο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας, για τη στήριξή σας τα προηγούμενα δέκα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Διαμαντούρο. Επόμενη ομιλήτρια εκ μέρου ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Επίτροπος Ρέντινγκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ καλό που σα ξαναβλέπουμε εδώ. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω όλο ιδιαίτερο τον κύριο Σαλαβράκο και την Επιτροπή Αναφορών για την εξαίρετη έκθεση που ετοίμασαν όσον αφορά τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Μεσολαβητή κατά το 2012. Η έκθεση αυτή είναι σημαντική γιατί μας δείχνει πόσο ελέγχεται εκείνους που ελέγχουν και βοηθήσατε έτσι πάρα πολύ τους πολίτες με το έργο που έλαβε χώρα όλα αυτά τα χρόνια. Και εσείς αναλάβατε αυτό το καθήκον και το κάνατε πάρα πολύ καλά κύριε Διαμαντούρο. Όλα αυτά τα χρόνια εσείς πρώτον οικοδομήσατε το θεσμό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και μετά ηγηθήκατε του θεσμού αυτού με υπομονή, με σοφία και επαγγελματισμό. Τα έχετε και τα τρία. Πιστεύω λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμπεριφέρθηκε σοφά τρεις φορές που σας ανέθεσε το καθήκον αυτό να ηγηθείτε του θεσμού του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Η έκθεση του κύριου Σαλαβράκου επίσης κάνει έναν απολογισμό και δείχνει τι επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια. Και φαίνεται ότι έγιναν συνεχώς προσπάθειες για να εμβαθυνθεί ο διάλογος με τους Ευρωπαίους πολίτες. Οι πολίτες πια γνωρίζουν ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Ευρωπαίου μεσολαβητή. Ο θεσμός αυτός λοιπόν γίνεται περισσότερο ορατός και αρχίζει να αποτελεί κομμάτι της καθημερινής ζωής των πολιτών. Αυτό είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Επίσης, Εμβαθύνοντας περισσότερο στο διάλογο όχι μόνο με τους πολίτες αλλά και με τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και με την κοινωνία των πολιτών, καταφέρατε να ενισχύσετε τα δικαιώματα των πολιτών και τη συμμετοχή τους στην δημοκρατική ζωή. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι χαίρουν μεγαλύτερες διαφάνειες και λαμβάνονται πιο υπεύθυνα. Αυτό είναι κάτι που χρειάζεται. Και αυτό το βλέπουμε, ιδιω τώρα το 2013, που είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών, βλέπουμε πως οι πολίτες ακόμα αγνοούν κάπως το πώς λειτουργούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αγνοούν το τι κάνει για αυτούς η Ευρώπη. Και ειλικρινά εξεπλάγει να πάνε ένα πρόσφατο ευρωβαρόμετρο που λέει ότι μόνο το 1 τρίτο των πολιτών πιστεύει ότι η φωνή τους ακούγεται και έχει κάποιο βάρος. Συνεπώς μένει πολλή δουλειά ακόμα να γίνει προκειμένου οι Ευρωπαίοι πολίτες τελικά να κατανοήσουν ότι ναι, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι για αυτούς, δουλεύουν για αυτούς και ότι εσείς κύριε Διαμαντούρο έχετε παίξει ζωτική σημασία ρόλο αλλάζοντας τις νοοτροπίες, τη διοικητική νοοτροπία και στρέφοντας την υπέρ των πολιτών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν γι' αυτό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις εξαιρετικές επιδόσεις που είχατε τα τελευταία αυτά δέκα χρόνια. Σας ευχαριστώ επίσης που τώρα στην ομιλία σας αναφερθήκατε και στις προκλήσεις για το μέλλον. Είπατε πώς εσείς βλέπετε αυτές τις μελλοντικέ προκλήσεις. Είπατε ότι συλλογικά πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε αυτές. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλω να πω ότι ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον κύριο Διαμαντούρο πάντα υπήρξε μια ανοιχτή σχέση με πίστη και αμοιβαίο σεβασμό. Συνεπώς για άλλη μια φορά κύριε Διαμαντούρο σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήσασταν εσείς που βρεθήκατε στο κέντρο αυτής της συνεργασίας. Σας εύχομαι λοιπόν και εγώ ό,τι καλύτερο για το μέλλον, υγεία και σίγουρα μία συνταξιοδότηση κατά τη διάρκεια της οποίας σίγουρα θα έχετε πολλές δραστηριότητες. Να ξέρετε ότι θα επανέλθω, δηλαδή επιτρέψτε μας να μπορούμε να στραφούμε σε εσά και στο μέλλον και να ζητήσουμε τις συμβουλές σας ξανά και ξανά, μια που μας βοηθήσατε τόσο πολύ αυτά τα τελευταία δέκα χρόνια. Κυρίες και κύριοι, τώρα για να έρθω πιο πολύ στα στοιχεία της σημερινής συζήτησης. Η έκθεση αναγνωρίζει τι τεράστιε προσπάθειες που έχουν κάνει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα γενικά, συμπεριλαμβανομένη και τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Υπάρχουν διάφορε καταγγελίες σχετικά με την διαφάνεια, αυξήθηκαν 36% το 2008 και 21% το 2012, κάτι το οποίο δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος και είναι πολύ ενθαρρυντική αυτή η τάση. Διαπίστωσε επίσης ότι οι περισσότερες από τις ε, έρευνες που έγιναν αφορούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και είναι λογικό αυτό, γιατί η Επιτροπή είναι και το κύριο θεσμικό όργανο της Ένωσης, το οποίο αποφάσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες. Διαπιστώνω όμως ότι ο αριθμός των ερευνών μειώθηκε το 2012 κατά 5%. Κάτι το οποίο δείχνει ότι ναι, μεν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αντικείμενο περισσότερων καταγγελιών, αλλά υπάρχει και μια φθήνουσα πορεία. Ίσως αυτό να συμβαίνει γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει σοβαρά υπόψη της και τις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητάει κοινού κανόνες και αρχές όσον αφορά τις διοικητικές διαδικασίες βάσει του άρθρου 298. Όχι, λάθος, 289 διορθώνει η κυρία Ρέντινγκ. Λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις λεπτομέρειες του διοικητικού δικαίου, όλες τις αδυναμίες και λήψεις που διαπιστώνονται στη διαχείριση των ευρωπαϊκών θεμάτων και όλα αυτά τα θέματα τα αναφέρουμε και στις χώρες μέλη. Στόχος μας είναι να συγκεντρώσουμε ό,τι πληροφορίες υπάρχουν όσον αφορά τα διοικητικά δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και να τα συγκεντρώσουμε σε μία ιστοσελίδα κεντρικά λίγο πολύ αυτό που υπογραμμίσατε κι εσείς κύριε Διαμαντούρο. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι πρέπει να ξέρουν πού πρέπει να απευθυνθούν και εκεί που απευθύνονται να έχουν και απάντηση. Αυτό είναι το βασικό για τα θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τα σχόλια του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή όσον αφορά την επέκταση του αεροδρομίου της Βιέννης και τις καταγγελίες που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση Δίας Πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να διευκρινιστεί το ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση για τροποποίηση της οδηγίας του 2011, την 92, όσον αφορά την ε, ε, αξιολόγηση τέτοιων προγραμμάτων σχετικών με το περιβάλλον. Είναι κάτι το οποίο στήριξε και η Επιτροπή Αναφορών και η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Οπότε τώρα αναμένω οι συνομοθέτες να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ τους και έτσι στο μέλλον να <coughs> μην χρειαστεί ειδική σύσταση από τη διαδοχό σας. Ο κύριος Αλαβράκος στην έκθεσή του υπογραμμίζει ότι σε 18 περίπου χρόνια ο διαμεσολαβητής έχει μόνο 18 ειδικέ εκθέσεις. Αυτό αποδεικνύει ότι πριν καταλήξουμε σε έκθεση από το διαμεσολαβητή έχει επιτευχθεί διακανονισμός, κάποια λύση το ότι μόνο σε 18 περιπτώσεις όλα αυτά τα χρόνια χρειάστηκε η ειδική έκθεση σημαίνει ότι έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, ότι επιτυχάνεται λύση πριν φτάσουμε σε αυτό το τελικό στάδιο. Πολύ θετικό. Αλλά για να διευκρινιστούν όλα αυτά τα ζητήματα και τα επερχόμενα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται με το ίδιο πνεύμα πίστης και επικοδομητικής συνεργασίας με την διάδοχό σας, την κυρία Έμιλι Ορέιλι, την οποία και συγχαίρω επί τη ευκαιρία για την εκλογή της. Προσβλέπω σε καλή συνεργασία μαζί της και αναμένω να τη συναντήσω. Στην Επιτροπή Αναφορών θέλω να πω επίσης ότι το έργο τους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έτος αυτών των πολιτών το είδα όταν είχα διάλογο με τους πολίτες, το διαπίστωσα ότι Πολλοί πολίτες γνωρίζουν την Επιτροπή Αναφορών. Και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν την ύπαρξή της οι πολίτες, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αυτό το οποίο εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες. Οπότε όταν κάτι δεν πάει καλά, είναι λογικό οι πολίτες πρώτα να σκεφτούν αυτούς που τους εκπροσωπούν και να απευθυνθούν σε αυτούς. Οπότε η συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή Αναφορών και τον διαμεσολαβητή λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Έτσι πρέπει να είναι. Και αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχουν σοφοί άνθρωποι και στην ε, Επιτροπή Αναφορών και είχαμε και έναν πάρα πολύ σοφό διαμεσολαβητή, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω για τα 10 χρόνια υπηρεσιών που μας προσέφερε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Επίτροπο. Φτάνουμε τώρα λοιπόν στους ομιλητές εκ μέρους των ε, πολιτικών ομάδων. Παρακαλώ να παραμείνετε στην, ε, ε, στο χρόνο ομιλίας σας και στην ημερήσια διάταξη. Για δύο λεπτά εκ μέρους του ΕΛΚ η κυρία Κολάρσκα Μπομπίνσκα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του ΕΛΚ θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον κύριο Διαμαντούρο για όλη την εργασία που κατάφερε να ολοκληρώσει τα τελευταία δέκα χρόνια η Επιτροπή των Αναφορών έχει συντάξει μία έκθεση η οποία δεν ήταν καθόλου αντιφατική. Όλοι συμφωνήσαμε ότι ήσασταν ένας εξαίρετος Ευρωπαίος ε, διομεσολαβητής κάνατε πιο διαφανή την ευρωπαϊκή διοίκηση και πιο αποτελεσματική. Από την άλλη όμως ε, έχετε εισαγάγει και κάποιες καινοτομίε, κάποιες αλλαγές. Μπορέσατε να βελτιώσετε την αντίδραση στις ε, προσφυγές των πολιτών. Στη διοίκηση δεν είναι πάντοτε δυνατό κανείς να αντιμετωπίζει θέματα περιεχομένου και καινοτομία. ταυτόχρονα. Εσείς τα καταφέρατε. Η δουλειά σας ε, το απέδειξε αυτό. Ως ε, ένα ενεργό μέλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων της Πολωνίας και αργότερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερα να ε, σας να, να δω πόσο εξαίρετο παράδειγμα διαμεσολαβητή ήσασταν. Το σύστημα αντίδρασης στις προσφυγές των πολιτών, στα αιτήματα των πολιτών και η γρήγορη έναρξη των ε, ερευνών ήταν πολύ σημαντική. Δώσατε επίσης ε, πολλές ε, χρήσιμες πληροφορίες στους πολίτες. Είναι σημαντικό οι πολίτες να κατανοούν τα δικαιώματά τους, την νομοθεσία και πώς λειτουργούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Ξεκινήσατε επίσης κατά πρωτοβουλία μια σειρά ερευνών, όπως ανέφερε και η Επίτροπος. προστατεύσατε τα συμφέροντα των πολιτών, όπως έγινε στην περίπτωση του αεροδρομίου της Βιέννης. Οι ευρωβουλευτές που είναι μέλη της Επιτροπής Αναφορών εκτιμούν τους κανόνες και το καταστατικό και τους κανόνες δεοντολογίας που θεσπίσατε. Αρχές όπως η αξιοπιστία, η οδετερότητα, η διαφάνεια ήταν χαρακτηριστικά σας. Δεν, μπορέσαμε, δεν μπορώ βέβαια να κατανομάσω όλα σας, τις, ε, όλα σας τα επιτεύγματα, αλλά ήσασταν ένας εξαίρετος ε, ε, διαμεσολαβητής. Ελπίζω ότι το ίδιο θα είναι και η κυρία Ωραίλη και θα συνεχίσει την παράδοση που εσείς ξεκινήσατε με τη θητεία σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρου τη ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για 1,5 λεπτό η κυρία Βέρτμαντ Αγγέλικα. Η κυρία Γκοντ Κίνκα. Ευχαριστώ κύριε ε, Πρόεδρε. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Διαμαντούρο εκ μέρους της ομάδας μας. Ε, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο διότι ήταν πάντοτε έτοιμος να δράσει και να παρέχει υπηρεσίες αλλά και διαφανείς υπηρεσίες. Ε, ήταν αμερόληπτος και υπήρξε μια καθόλου σεβαστή προσωπικότητα. Εδώ και δέκα χρόνια ο κύριος ε, Διαμαντούρος ήταν ε, ένας ε, εξαίρετος Ευρωπαίος διαμεσολαβητής. Είχαμε χιλιάδες προσφυγές πολιτών αλλά και αιτήματα για πληροφορίες τα οποία αντιμετώπισε σχετικά με θέματα που αφορούσαν τους πολίτες. Ήτανε πολύ καλός Ευρωπαίος ε, διαμεσολαβητής ε, σε όλα αυτά τα καθήκοντα. Μέσα σε αυτά τα δέκα χρόνια ε, μειώθηκε το ποσοστό των πολιτών που ζητούν πληροφορίες. Αυτό δείχνει ότι οι πολίτες πια παίρνουν πληροφορίες μέσα από τον διαδικτυακό τόπο. Οι ευρωβουλευτές ε, θέλαμε επίσης να έχουμε ένα άμεσο σύνδεσμο με την ε, ιστοσελίδα σας έτσι ώστε να σας βοηθήσουμε στη δουλειά σας και να μας βοηθήσετε. Ε, επίσης υπήρξε μεγάλη υποστήριξη από την πλευρά σας στα άτομα με αναπηρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η, συμφωνία του, η Σύμβαση του ΟΗΕ προσχώρησε τη συμφωνία του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρία, αναπηρία με βάση τις δικές σας συστάσεις. Ελπίζουμε ότι και η επόμενη Ευρωπαίος Διομεσολαβητής ε, θα τηρήσει τις ίδιες αρχές και θα διασφαλίσει για τα άτομα με αναπηρία τα ίδια δικαιώματα. Για παράδειγμα για τους ε, τυφλούς. Ε, εδώ πέρα, χθες σε ευρωπαϊκό επίπεδο είχαμε ένα πολύ καλό παράδειγμα για το τι συμβαίνει με τα άτομα με αναπηρία. Ευχαριστούμε πολύ. Για 1,5 λεπτό, εκ μέρου ε, του Άλντε, η κυρία Βέρτμαν Αγγέλικα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Αντιπρόεδρε, κύριε Διαμαντούρο. Δέκα χρόνια πέρασαν και ε, φαίνεται ε, σε όλους μας πια ξεκάθαρα πόσο καλή δουλειά έχει κάνει ο κύριος Διαμαντούρος. Να τονίσω την διαφάνεια παρόλο που δεν υπάρχει μεγάλη διαφάνεια ε, στην ε, ε, εργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται υπάρχει μάλλον, φαίνεται ότι οι πολίτες δεν αισθανόταν ακριβώς το ίδιο. Έτσι λοιπόν βοηθήσατε στο να δοθούν πληροφορίες στους πολίτες. Υπήρχαν λοιπόν όργανα, ιδρύματα και διάφορες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες κατάφεραν να συνεργαστούν καλά με τον διαμεσολαβητή, να διασφαλίσουν έτσι μια βελτίωση της εικόνας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, το αεροδρόμιο στη Βιέννη δείχνει ε, πόσο καλά συνεργάστηκαν όλοι οι συμμετέχοντες. Μπορέσατε να βρείτε καλή λύση για όλους. Τέλος, εγώ ως εισηγητρία για την έκθεση για τις γυναίκες με αναπηρία να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε και στις ανάγκες των πολιτών τις οποίες φροντίσατε ε, με πολύ μεγάλη προσοχή. Όπως υπόθηκε, ε, αναφέρω, υπο, περιλαμβάνω σε αυτούς ε, όχι μόνο τα άτομα με αναπηρία αλλά και τα παιδιά και ε, το γεγονός ότι προσχωρήσαμε στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα για την, με αναπηρία και σας ευχαριστούμε πολύ για όλη σας αυτή τη συμβολή. Ευχαριστούμε πολύ τη συνάδελφο. Ο συνάδελφος Ρούμπριχ, έχετε κάποια ερώτηση? Ζητάει το λόγο. Ναι, σωστά. Θα ήθελα να ρωτήσω τη συνάδελφο Βέρτμαν. Ε, για μας όλους η διαφάνεια είναι πολύ σημαντική και ο, ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής ε, το έχει ε, κάνει αυτό πραγματικότητα. Ξέρετε ότι υπάρχει ένας κατάλογος για τους όσους ασκούν πίεση υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις διότι βλέπουμε ποια είναι τα συμφέροντα που εκπροσωπούν και πώς χρηματοδοτούνται από την Ευρώπη. Παρακαλώ. Αγαπητέ συνάδελφε Ρούμπικ, και εγώ συμφωνώ ε, και νομίζω ότι θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα στον τομέα της διαφάνειας. Ε, θεωρώ ότι και η διάδοχος του κυρίου Διαμαντούρου θα δεσμευτεί και θα εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση και θα διασφαλίσω ώστε η αντίστοιχη επιτροπή να πέσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε την συνάδελφο. Για δύο λεπτά δίνω το λόγο στην ε, κυρία Όκεν εκ μέρους ε, των Πρασίνων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω τρία πράγματα που θέλω να πω. Καταρχάς, ε, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Σαλαβράκο για την εξαίρετη έκθεσή του και μετά ένα ε, μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Διαμαντούρο για την εξαίρετη εργασία του που έχει συμβάλει στο να γίνει ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ένας πάγιος θεσμός. Δεν ξέρω αν είναι πλήρως πάγιος, αλλά ελπίζω ότι ε, μετά από 10 χρόνια ε, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Είναι ένας θεσμός στον οποίο μπορούν να προσφύγουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και σας ευχαριστώ επίσης γιατί ε, φαίνεται ότι μια παράδοση συνεχίζεται και παρά τις δυσκολίες έχουμε έναν πραγματικό διαμεσολαβητή που συνεχίζει να χτίζει πάνω στις βάσεις που έχουν τεθεί. Ελπίζω λοιπόν ότι θα υπάρχει αυτή η εγγύηση για τους πολίτες ότι θα έχουν καλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αναφερθώ επίσης στη συνεχή ε, στις έλλειψη νομοθεσίας και κανονισμών για την καλή διαχείριση να ζητήσω από την Επίτροπο Ρέντινγκ να φροντίσει αυτό το θέμα, να τεθούν τα συμφέροντα των πολιτών ε, σε πρώτη μοίρα σε σχέση με αυτά των ε, αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίζει ότι οι πολίτες αντιμετωπίζονται σωστά και κατανοώ ότι είναι πολλές φορές δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Κάτι τελευταίο που ήθελα να αναφέρω είναι κάτι που ανέφεραν και όλοι οι υποψήφοι για τη θέση του διαμεσολαβητή. Ότι θα πρέπει ε, να υπάρχει διαφάνεια και ε, στην βιομηχανία την ιατρική το γεγονός ότι έχει ε, παρέμβει το δικαστήριο έχει παραλύσει τα πράγματα εδώ και δύο χρόνια και είναι σκάνδαλο που ε, παραγωνίζεται η απόφαση του Ομπούτσμαν, η απόφαση η δική μας, η χάρτα. Τι θα γινόταν αν κέρδιζε η βιομηχανία, τι θα γινόταν με την υγεία των πολιτών. Σας ευχαριστούμε λοιπόν κύριε Διαμαντούρε για την εξαίρετη δουλειά σας Ευχαριστούμε την συνάδελφο. Επόμενος ομιλητή για 1,5 λεπτό και πάλι εκ μέρους ε, τη ΓΚΟΕ, ο κύριος Χουντή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρου τη ομάδα τη Ενωτική Αριστερά ε, θέλω να πω ότι υποστηρίζουμε την έκθεση του συναδέλφου του κυρίου Σαλαβράκου, άλλωστε έχει την καθολική υποστήριξη στην Επιτροπή Αναφορών και βεβαίω αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι αποτιμά θετικά το έργο του ευρωπαίου διαμεσολαβητή. επιτρέψτε μου λοιπόν κύριε πρόεδρε εκ μέρου τη ενωτική αριστερά τη ομάδα να ευχαριστήσουμε και εμεί τον κύριο διαμαντούρο για αυτή τη δεκαετή προσφορά στο λειτουργήμα του ευρωπαίου διαμεσολαβητή. έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά έχει την καθολική αναγνώριση και έκανε τη δουλειά του πολλέ φορέ μέσα σε δυσκολίε και όχι σε διευκολύνσει από τα όργανα τη ευρωπαϊκή ένωση και κυρίως κατά την άποψή μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να κάνω λοιπόν μια γενικότερη παρατήρηση για τη ε, δράση και τη δουλειά του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή που βεβαίως ισχύουν για την νέα που ανέλαβε ε, το λειτουργήμα αυτό. Αυτό που πρέπει για να γίνεται πολύ αποτελεσματική η δουλειά χρειάζεται να έχει τη δυνατή βοήθεια όλων των θεσμών και όλων των οργάνων του ευρωπαϊκού οικοδομήματος το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και με τη σημερινή συζήτηση εκφράζει την υποστήριξη στη δουλειά του ευρωπαίου διαμεσολαβητή. αυτό πρέπει να το κάνουν και τα άλλα όργανα. το δεύτερο που θέλω να πω λόγω τη κρίση η οποία σοβεί ιδιαίτερα στι χώρε του νότου είναι σίγουρο ότι πολλά προβλήματα θα εμφανιστούν υπό τη μορφή κακοδίκηση και θα ενταχθούν στο αντικείμενο του ευρωπαίου διαμεσολαβητή. κατόπιν τούτου είναι πάρα πολύ κρίσιμο εκτό των άλλων να λειτουργούν τα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια, ούτω ώστε οι πολίτε να έχουν ένα αποκούμπι στη δουλειά του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, σε αιτήματα που ε, διατυπώνουν και σε αδικία που γίνεται σε βάρο του να μπορούν να βρίσκουν το δίκαιο του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο. επόμενο ομιλητή για 1,5 λεπτό μέρους ε, της Ευρώπης της και της ο κύριο Πάσχα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Διαμεσολαβητή. Η ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2012 συνοψίζει τις ε, επιδόσεις αυτής ε, της υπηρεσίας τα τελευταία 10 χρόνια στην ουσία. Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετούς θητείας του ο κύριος Διαμαντούρος έχει εκτελέσει εξαιρέτως τα, του και τα καθήκοντά του και έχει δημιουργήσει μια υπηρεσία η οποία δικαιώνει τον διαμεσολαβητή και την Ένωση. Σε επίπεδο στατιστικών είναι πολύ σημαντικό να διαπιστώσουμε ότι χάρη στην ε, εκστρατεία πληροφόρηση του διαμεσολαβητή, οι πολίτες κατάφεραν να κατανοήσουν την κατανομή δυνάμεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Η προστασία των πολιτών είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της ευνομούμενη κοινωνίας. Βλέπουμε στην ουσία πώς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χρησιμοποιούν τις βέλτιστες πρακτικές, γιατί ε, ε, υπήρξε μεγάλη ε, αύξηση στις έρευνες ε, για τις παραβιάσεις δικαιωμάτων και από το Κοινοβούλιο και από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα γενικότερα. Επίσης, διασφάλισε τις καλές σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Για να καταλήξω θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για την εξαίρετη εργασία του ως Διαμεσολαβητή και να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την εξαίρετη δουλειά που έκανε κατά τη σύνταξη της, ε, προ... της έκθεσης που συνοψίζει τα όσα υπόθηκαν στην Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Φλαζάκ, ε, το ECR. Vážený pane předsedo, dámy a Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η δουλειά του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και ήταν μεγάλη σημασία στα τελευταία χρόνια και εκ μέρους της ομάδας μου θα ήθελα να τον ευχαριστήσω. Να μην ξεχάσουμε όμως ότι υπάρχει ακόμα χώρος για βελτιώσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι τα δικαστήρια έχουν το δικαίωμα ε, να ε, λαμβάνουν δεσμευτικές αποφάσεις. Η θητεία του διαμεσολαβητή στην ουσία σχετίζεται με συστάσεις και έρευνες ο διαμεσολαβητής ε, μπορεί να αντιδράσει βελτιώνοντας την ποιότητα ε, και διασφαλίζοντας την ηθικότητα. Υπάρχει όμως, όπως είπα, χώρος ε, για βελτίωση και γι' αυτό θα θέλαμε να προσκαλέσουμε τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να διαβάσει τις διάφορες εκθέσεις και να δει που έκανε λάθος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουν ε, ε, γίνει πολλές προσφυγές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πραγματικά πρέπει να ληφθούν μέτρα για να βελτιωθεί η δράση του. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί η χρήση των κατάλληλων μέσων που χρησιμοποιούνται ε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Πολλές ε, ε, φορές ε, επίσης θα πρέπει να αναφέρ... Θα πρέπει επίσης να αναφερθούμε και στο κόστος της επίλυσης των διαφορών. 13.000 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 13.000 κορώνες στην Τσεχία. Αυτό πραγματικά επιβαρύνει πολύ τον προϋπολογισμό. Παρόλα αυτά, αυτό ισοσταθμίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη δουλειά σε εθνικό επίπεδο. Στις επόμενες ε, εκθέσεις των επόμενων ετών ε, πιστεύω ότι ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να αντιμετωπίσει τέτοια θέματα. Ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στον επόμενο μιλητή. Για δύο λεπτά έχει το λόγο ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκεστε και πάλι μαζί μας αγαπητέ κύριε Διαμαντούρο. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε ότι ο Ευρωπαίος Διαμασελαβητής ο κύριος Διαμαντούρος έκανε και το 2012 μια πολύ καλή δουλειά. Είχαμε χιλιάδες, δεκάδες ε, προσφυγές τις οποίες αντιμετώπισε θα έγιναν διάφορες έρευνες ε, οι οποίες ε, παρουσίασαν αύξηση κατά 18% σε σχέση με το παρελθόν και πραγματικά υπήρχε ε, και το θέμα του αεροδρομίου που ήταν ένα το παράδειγμα της καλής συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Βλέπουμε ότι χιλιάδες πολίτες μπόρεσαν να βρουν άμεσα βοήθεια και αυτό είναι ένα πολύ ευχάριστο αποτέλεσμα. Βασικές αρχές ε, της ευρωπαϊκής ε, διοίκησης όπως η ακαιρεότητα, αντιμεκειμενικότητα, ο σεβασμός των άλλων, η διαφάνεια ήταν αρχές ε, που εκπροσωπούσε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Αρχές που πρέπει να τηρεί ο καθένας από εμά και ο Ευρωβουλευτής και ως άνθρωπος. Επίσης υπάρχει και ο Ευρωπαϊκός Κώδικας για καλές ε, διοικητικές πρακτικές ε, που προωθήθηκε με τη βοήθειά του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Διαμαντούρο για τη δουλειά του το 2012 και για την ε, ιδιαίτερη δέσμευση που επέδειξε τα τελευταία 10 χρόνια. Δημιούργησε ένα αποτελεσματικό δίκτυο Ευρωπαίων Διαμεσολαβητών και βοήθησε χιλιάδες πολίτες. Μπόρεσε να κάνει τη διοίκηση πιο αποτελεσματική και διαφανή και έχει διαμορφώσει το τοπίο ε, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Επίσης υπάρχει χώρος ε, για βελτίωση, να βελτιωθεί ας πούμε συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Αναφορών και των Ευρωπαίων Διαμεσολαβητών. Παρόλα αυτά το δικό σας έργο, αυτό που αφήνετε πίσω είναι πραγματικά αξιοσημείωτο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο. Εκ μέρους... Ε, ε, επόμενη ομιλήτρια για δύο λεπτά η κυρία Μποστινάρου. Κύριε Πρόεδρε, ε, καλωσορίσατε ορίσατε και πάλι. Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Διαμεσολαβητή, κύριε Διαμαντούρο θα έλεγα ότι είναι μάλλον ξεχωριστό το να ακούσουμε ομιλητές από όλες τις ομάδες να μιλάνε με τον καλύτερο τρόπο, στον υπερθετικό βαθμό για τον θεσμό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Αυτό, αυτός είναι ο φόρος τιμής που αποτεί το Κοινοβούλιο στον κύριο Νικηφόρο Διαμαντούρο μετά από 10 χρόνια ε, θητείας. Αγαπητέ φίλε Νικηφόρε, σε ευχαριστούμε που υπήρξες πάντοτε διαθέσιος, σε ευχαριστούμε που συνέβη στο να προωθηθεί η διαφάνεια και η κουλτούρα της καλής διοίκησης, ε, της χρηστής διοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τον διακεκριμένο τρόπο με τον οποίο έδρασε στα 10 χρόνια. Ένας από τους πιο επιτυχημένους φακέλους του 2012 ήταν αυτός που αφορούσε το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βιέννης. Ε, μια θαυμάσια συνεργασία η οποία κατέληξε σε μια ομόφωνη ψηφοφορία και που επέτρεψε την Επιτροπή Επιτροπή ε, Αναφορών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρουν λύσεις για το μέλλον. Αυτή η έκθεση μας έδωσε τη δυνατότητα να συμβάλλουμε με τη σειρά μας στην τροποποίηση του σχεδίου οδηγίας που αφορούσε την επίπτωση του εδρομίου στο περιβάλλον έτσι ώστε τα πράγματα αυτά δεν θα επανεληφθούν στο μέλλον. Δεν μπορώ παρά να καλωσορίσω την έκθεση Ζανόνη η οποία έλκει την έμπνευσή της ε, μεταξύ των άλλων από τις ε, δραστηριότητες της Επιτροπής ε, Αναφορών. 52,7% των ερευνών του 2012 που ξεκίνησαν από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή είχαν στόχο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη της ότι υπάρχει περιθώριο για καλύτερη διοίκηση σε αυτό το επίπεδο. Τα πρότυπα που έχετε θέσει είναι τα πρώτα τύπα στα οποία θα βασιστεί η νέα διαμεσολαβήτρια και είμαι πεπισμένος ότι η δραστηριότητα της κυρίας Ορέλη θα σταθεί στο ύψος αυτών των ποιοτύπων. Ε, στο επαντή κύριε Διαμαντούρο και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να σας θυμίσω ότι είναι λίγο φιλόδοξη η μερίσια διάταξη. Παρακαλώ να παραμείνετε πιστοί στο χρόνο ομιλία σας. Είμαι αισιόδοξο ότι η συνάδελφος ε, Γετλιμέκη θα χρησιμοποιήσει καλά το χρόνο της. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε, χαίρομαι και πάλι που σας βλέπω να καταλαμβάνετε τη θέση σας και να είστε και τόσο καλά μεταξύ των άλλων. Κύριε Διαμεσολαβητή, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα πεπραγμένα σας πραγματικά. Τα όσα κάνατε ήταν πολύτιμα και σε, ε, κάτω από συνθήκες όχι πάντοτε εύκολες. Προωθήσατε την ιδέα της διαφάνειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθήσατε την ιδέα της καλής διαχείρισης, προωθήσατε μία σειρά από αξίες ενώ πολλοί εναντιώθηκαν σε αυτό και καταφέρατε εξαίρετα αποτελέσματα. Η κρίση των τελευταίων ετών απεκάλυψε ότι υπάρχουν κενά ως προς τη διαφάνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν προβλήματα με τις τράπεζες προβλήματα οποία συγκαλύφθηκαν από τις χώρες μέλη, κάτι που οδήγησε σε μία ενδυνάμωση της κρίσης. Θα πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε μια προσπάθεια έτσι ώστε να μην επαναληφθούν όλα αυτά. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τη διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα επίπεδα γιατί αυτό καλλιεργεί την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτή τη φορά δεν το καταφέραμε. Χρειαζόμαστε κανονισμούς που να αφορούν τις βέλτιστες διοικητικές πρακτικές. Είμαι σίγουρη ότι εσείς τα κάνατε όλα αυτά κατά τη διάρκεια της εντολής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαίρετη, το εξαίρετο που επιτελέσατε. Σε περίπτωση που έχετε δει τον ε, κύριο Χέλμερ, γιατί εγώ δεν τον βλέπω, αν τον βλέπετε εσείς ε, πείτε μου, αλλιώς ε, πάμε στην επόμενη ομιλήτρια. Για δύο λεπτά η κυρία Ματζόνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχές και από μένα καλώς ορίσατε και πάλι. Καλώς επανήλθετε. Η ε, ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, όπως ακούσαμε, αποτελεί και έναν απολογισμό του τέλους της θητείας του. Ο φίλος κ. Διαμαντούρος αποφάσισε να διακόψει την ε, πορεία του πριν από το τέλος της θητείας του. Συνεπώς ε, κλείνει μία δεκαετία με έναν απολογισμό δίχως άλλο εξαιρετικό. Τα στοιχεία που αφορούν την αποτελεσματικότητα, την ικανοποίηση των πολιτών αποτελούν μαρτυρία της δέσμευσης του κυρίου Διαμαντούρου, ο οποίος κατάφερε να επενδύσει αυτά τα χρόνια και να συμβάλλει στην προώθηση μία καλύτερης σχέσης με το μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων του διαμεσολαβητή και των ε, πολιτών. Ως πρόεδρος ε, της Επιτροπής Αναφορών θα ήθελα να τονίσω ότι βελτιώθηκε η σχέση μεταξύ του διαμεσολαβητή και της ίδιας της Επιτροπής. Αυτή η αποδοτική συνεργασία έδειξε ότι το δίκτυο αυτό λειτουργεί και ότι αποτελεί ένα πάρα πολύ έγκυνο εργαλείο. Αυτό συμβάλλει στην εδραίωση μιας σχέσης μεταξύ ε, πολιτών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ε, με αυτόν τον τρόπο προφυλάσσεται ο σεβασμός <coughs> των θεσμών κατά τους πολίτες η λειτουργία αυτή είναι σημαντική και χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι ευγνώμος στον κύριο Διαμαντούρο ο οποίος προήγαγε αυτή την αντίληψη. Ευχαριστούμε πολύ την συνάδελφο. Επόμενος ομιλη... Ε, επόμενη ομιλήτρια η κυρία Γκέριγκερ Ντε Όντενμπεργκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με λύπη άκουσα ότι ο καθηγητής Διαμαντούρος δεν θα είναι πλέον Ευρωπαίος διαμεσολαβητής γιατί την τελευταία δεκαετία εργάστηκε πραγματικά <coughs> με αξιοθαύμαστο τρόπο ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την διαφάνεια των διαδικασιών και την παροχή καλύτερων πληροφοριών στους πολίτες. Τα τελευταία χρόνια ποιήσε πάνω από 2.500 καταγγελίες που αφορούσαν κακή διοίκηση. Παρήχε στοιχεία για πάνω από 20.000 περιπτώσεις. Αν κοιτάξετε τον αριθμό των ερευνών θα διαπιστώσετε ότι υπήρξε μία αύξηση κατά 23% σε σχέση με το 2011. Το... Οι αιτήσει για παροχή πληροφοριών ε, ε, μειώθηκε, το οποίο σημαίνει ότι η διαδραστική στο σελίδα που ε, δημοσι... υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματική. Επίσης, ο αριθμός των καταγγελιών δεν ανήκουν στην ε, έφτασε το χαμηλότερο επίπεδο την προηγούμενη χρονιά. Παρόλα αυτά η έκθεση μας δείχνει ότι η πρόσβαση στα <clears throat> έγγραφα και η διαφάνεια ορισμένων διαδικασιών δεν είναι επαρκή. Το, 22, ε, ε, το κλείσιμο 22% των περιτόχων έχουν σχέση με αυτό. Υπήρξε και μία αύξηση το μέσο αριθμό αναμονής για να ξεκινήσει μια διαδικασία. Ανακεφαλαιώνοντας, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τα επιτεύγματα των τελευταίων ετών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που εργαστήκατε προάγοντας <clears throat> τη χρηστή διοίκηση. Θα ήθελα να σας ευχηθώ ό,τι, καλύτερα, ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ τη συνάδελφο. Επόμενη μιλήτρια για ένα λεπτό η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω τη δυνατότητα να σας καλωσορίσω. Χαίρομαι επίσης που μου δίνετε τη δυνατότητα να ευχαριστήσω τον διαμεσολογητή κύριο Διαμαντούρο για τα όσα επετέλεσε των όμετος ε, ε, προς όφελος των Ευρωπαίων ε, πολιτών. Καταφέρατε να δράσετε με ένα αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο. Νομίζω ότι το γραφείο του διαμεσολαβητή βρέθηκε σε καλά χέρια. Καταφέρετε να γεφυρώσετε το κενό του δημοκρατικού ελλείμματο μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Χαίρομαι που μία από τι προτεραιότητέ σα ήταν να διατηρήσετε το διάλογο. Η εμπλοκή των ανθρώπων ε, ε, σε επίπεδο ευρωπαϊκό δεν περιορίζεται μόνο στην περίοδο των εκλογών. Ο πολίτη βρίσκεται αντιμέτωπο με πάρα πολλά εμπόδια, αποθαρρύνεται, χάνει την εμπιστοσύνη του. Νομίζω ότι εσεί, συμβάλλατε στο να καταστήσετε απλή αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελα να ευχηθώ ότι καλύτερο στη νέα διαμεσολαβήτρια, την κυρία Οράιλι. δίχω άλλο θα βρεθείτε μπροστά σε καινούριε προκλήσει, αλλά η δέσμευση είναι το σημαντικό για να μπορέσετε Έστε επιτελέσετε σωστά το ρόλο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Κέλλη για δύο λεπτά. Ε, uh, κύριος Κέλλη. Ε, θα έλεγα ότι δεν είναι σύνηθες το να υπάρχει απόλυτη ομοφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα ε, βρισκόμαστε μπροστά σε μία εξαίρεση. Κυρίως γιατί ο διαμεσολαβητής, ε, κύριος Διαμαντούρος, ε, αφοσιώθηκε σε αυτό που έκανε τα τελευταία δέκα χρόνια. Δεν δούλεψε μόνο με επαγγελματισμό αλλά και με σοφία, με υπομονή. Πραγματικά συνειδητοποιώ ότι εσείς είστε ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτή την εργασία. Γιατί δεν έχετε να υπερεγω. Εσείς θέλατε να παράσχετε τις υπηρεσίες σας και αυτό είναι μια σωστή αντίληψη. Ε, τις θερμότερες ευχές μου και θα ήθελα να ευχηθώ και στην κυρία Ορέιλι, τη συμπολίτησά μου, ό,τι καλύτερο στο νέο έργο που ανέλαβε. Πιστεύω ότι κύριε ε, Διαμαντούρο μπορείτε να είστε πάρα πολύ περήφανος για το έργο που επιτελέσατε. Πολύ συχνά η γραβιοκρατία απογοητεύει τους πολίτες Χαίρομαι που υπάρχει αυτός ο φορέας που συγκεντρώνει τις καταγγελίες των πολιτών. Εκτός από αυτό, εσείς καταφέρατε να βοηθήσετε 22.000 άτομα. Τα συμβουλέψατε, τους είπατε τι να κάνουν και συμβάλλατε στο να καλυφθεί, να γεφυρωθεί αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα που υπάρχει. Κάτι άλλο σημαντικό. Ο διαμεσολαβητής διατυπώνει παρατηρήσεις όταν ε, υπάρχουν καταγγελίες ενώ στο παρελθόν ε, εάν ο πολίτης δεν ικανοποιεί ε, ε, κατήγγειλε και πάλι το σύμβαν. Εσείς καταφέρατε να βοηθήσετε τους πολίτες. Ευχαριστούμε λοιπόν. Ειδικότερα από την πλευρά μου ε, να σας ευχαριστήσω γιατί πραγματικά ήσασταν ο μοναδικός που τήρησε το χρόνο του σήμερα. Για ένα μισή λεπτό ο κύριος Κάσμαν. Thank you very much, President. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος... Τι να πω κύριε Διαμαντούρο, ακούγοντας ε, τα Όσα ακούσατε σήμερα ήταν σαν να είναι μια νεκρολογία, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Είναι καταπληκτικό αυτό που κάνατε. Ε, μας βοηθήσατε να έχουμε πρόσβαση σε έγγραφα. Είναι κρίμα που πολλές από τις καταγγελίες αφορούν την ε, ε, πρόσβαση στα έγγραφα και την διαφάνεια. Εσείς φροντίσατε έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη λογοδοσία των ε, θεσμικών οργάνων προς τους πολίτες Κάνατε πάρα πολλά για τους ε, ανάπηρους. Πραγματικά μας ε, βοηθήσατε με έναν τρόπο που δεν θα μπορέσουμε να ξεχάσουμε. Θα θέλω να πω επίσης ότι το γεγονός ότι η Έμιλι Οράιλι θα είναι η η επόμενη διαμεσολαβήτρια μας θυμίζει ότι θα πρέπει να είναι πολιτικά ε, ουδέτερη. Ναι, θα φύγετε, ναι, η θητεία σας εδίρκεσε δέκα χρόνια και ήταν καταπληκτική. Εμείς θα ακολουθήσουμε την δική σας γραμμή, εμείς την Επιτροπή Αναφορών Υπάρχουν θέματα που δεν έχουν επιληθεί, αλλά κύριε Διαμαντούρο, ξέρουμε ότι το πάθος σας θα παραμείνει και πιστεύω ότι ένα από τα καλύτερα πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι η δική σας κληρονομιά θα διασφαλίσει το δρόμο που θα ακολουθήσει η κυρία Ορέιλι. Ευχαριστούμε πολύ αγαπητές συνάδελφοι. Επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό, ο κύριος Κάτσακ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, κύριε Διαμαντούρο, Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω από βάθος καρδίας για όλες τις προσπάθειες που κάνατε μέχρι τώρα και για όσα καταφέρατε στον τομέα της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φροντίσατε επίσης για την εξέλιξη του θεσμού αυτού, του διαμεσολαβητή, προκειμένου να εγκαθιδρυθεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 67% των καταγγελιών έγιναν μέσω διαδικτύου. Πολύ σημαντικό λοιπόν το ότι υπάρχει στο σελίδα σας αυτή. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές καταγγελίες σχετικά με τη διαφάνεια των ευρωπαϊκών θεσμών οι καταγγελίε αυτέ, ο αριθμό δηλαδή των καταγγελιών αυτών είναι σχετικό γιατί δείχνει τη δυσπιστία των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Γι' αυτό λοιπόν και κάνω έκκληση στην κυρία Ορέιλι που θα σα διαδεχθεί να συνεχίσει το έργο σα ώστε να τεθεί ο πύχη τη διαφάνεια όσο γίνεται πιο ψηλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο ο ο κύριος Μπέκερ για δύο λεπτά. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμε κύριε Διαμασολαβητή, αγαπητοί συνάδελφοι, για τον απολογισμό το 2012 αλλά και για όλη σας τη θητεία θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Διαμαντούρο γιατί πραγματικά ήσασταν ιδιαίτερα επαγγελματίας και ένας εταίρος της Επιτροπής Αναφορών ως Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Εγώ ε, θα ήθελα να αναφερθώ ειδικότερα στην έκθεση για το αεροδρόμιο της Βιέννης ε, και τις επιπτώσεις που είχε. Οδήγησε σε βελτίωση των διαδικασιών και μία διεύρυνση ε, των τρόπων με τον οποίο μπορεί να εκφράζεται η Κομισιόν. Έχουμε μια πιο αποτελεσματική συμμετοχή του κοινού όπως είδαμε επίσης και τον Οκτώβριο στην αναθεώρηση της σχετικής οδηγίας. Ε, ε, μάθαμε λοιπόν να δουλεύουμε πιο αποτελεσματικά. Αναγνωρίζω πραγματικά ε, σε όλους τους διαμεσολαβητές ικανότητες, προσωπική δέσμευση. Ελπίζω ότι προνόμια όπως η στοχοθεσία, η επικοινωνιακή εργασία και η εντατική χρήση του online οργάνου που θα οδηγήσει ώστε να μπορούν οι πολίτες να παρακολουθούν τις αιτήσει τους ε, online ε, θα συνεχίσουν. Επίσης, ε, να συνεχίσει η εργασία, η ποιοτική εργασία που έχουμε επιτύχει με τον κύριο Διαμαντούρο στην Επιτροπή Αναφορών και με τους επόμενους υπόλοιπους διαμεσολαβητές. Εμείς ε, εξυπηρετούμε τους πολίτες της Ευρώπης. Ε, σας εύχομαι εκ μέρους αυτών και ε, εμού, εμού προσωπική υγεία και ευτυχία στην προσωπική σας ζωή. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Έρτουπ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ξαναβλέπω εδώ. Mm. Κύριε Διαμαντούρο, σας ε, εύχομαι ό,τι καλύτερο για την υπόλοιπη ζωή σας και σας ευχαριστώ για τα 10 χρόνια που εργαστήκατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τελευταία δημοσκόπηση έδειξε ότι το 10% των πολιτών ε, θεωρεί ότι ο Ευρωπαίος Διαμοσολαβητής ε, έχει ε, ως καθήκον να προωθεί τα αιτήματά τους και να τους δίνει πληροφορίες. Είναι μια πρόοδος, αλλά είναι μικρό το ποσοστό ακόμα. Μπορούμε περισσότερα να κάνουμε. Έχουμε μισό δις κατοίκους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν έχω κάνει σωστά την έρευνα το 2012... Έχουμε 2.450 περίπου καταγγελίες ε, ήταν λίγες. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι ενημερωμένοι επαρκώς οι πολίτες. Θεωρώ όμως παρόλα αυτά ότι το 14% των πολιτών που θεωρούν ε, ότι δεν είναι διαφανής η Ευρωπαϊκή Ένωση μας δείχνει πόση δουλειά μπορεί να γίνει ακόμα. Σας ευχαριστούμε όμως για τη δουλειά σας κύριε Διαμαντούρα. Ευχαριστούμε. Ο επόμενος ομιλητής... Ο κύριος Ιρτουγκάη Άγγουλο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ετήσια έκθεση για τι δραστηριότητε του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2012 είναι ιδιαίτερη γιατί λαμβάνει χώρα τώρα που γνωρίζουμε ότι θα μα εγκαταλείψει ο κύριο Διαμαντούρο. Τα επιτεύγματα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι τεράστια. Τον ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που προώθησε μια νοοτροπία καλή εξυπηρέτηση και χρηστή διοίκηση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Επίσης τον ευχαριστούμε πολύ για την τόσο καλή συνεργασία που είχε με την Επιτροπή μας Αναφορών. Θέλω να συγχαρώ και τον φίλο μου τον κύριο Σαλαβράκο για την δικιά του έκθεση, για το εξαίρετο έργο του προκειμένου να εκπονήσει την έκθεση αυτή. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι υπάρχουν πολλά θετικά, κύριε Πρόεδρε, που έχουν να κάνουν με τι δραστηριότητε του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2012. Και κυρίω τα εξή. Το γεγονό ότι το 67% των καταγγελιών υποβλήθηκε διαδικτυακά κάτι το οποίο δείχνει ότι ο θεσμός του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή προσαρμόζεται στις επιταγές της εποχής μας. Έπειτα ότι υπάρχει ε, διάδραση. Είναι πολύ σημαντικό. Κάθε φορά που φτάνουν καταγγελίες από τους πολίτες, χάρη στο διαδίκτυο, μπορούν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη των καταγγελιών τους οι πολίτες είναι πολύ σημαντικά, όπως επίσης η νέα εκδοχή του κώδικα διοντολογίας. Είναι πολύ σημαντικό γιατί συμπεριλαμβάνει τις αρχές της χρηστής ε, ε, δίκησης και λαμβάνει την υπόψη από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Το τρίτο, το πολύ σημαντικό, είναι το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων για το οποίο αφιέρωσε ιδιαίτερη πρόσοχη το 2012 Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, όπως επίσης και η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες, τα δικαιώματά τους. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ε, λαμβάνουμε υπόψη μας τα δικαιώματα αυτά και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στη Σύμβαση των ΗΠΑ για τα δικαιώματα των ατόμων αυτών με αναπηρία. Επίσης πολύ σημαντικό είναι το θέμα της συνεργασίας με ολόκληρο το δίκτυο των ε, διαμεσολαβητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο πιστεύω τελικά ενισχύει τη διαφάνεια των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν τον κύριο Σαλαφράκο εκ μέρου του ΕΡΚ που ανέλαβε την έκθεση αυτή και ευχαριστώ πολύ για το έργο σα κύριε Διαμαντούρο. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο. Για ένα λεπτό ο κύριος Μύρισκη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Διάβασα με ιδιαίτερη προσοχή την έκθεση που αφορά τις δραστηριότητε σα, κύριε Διαμεσολαβητά, και ευχαριστώ πολύ. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει ένα έργο το οποίο δεν ολοκληρώσατε. Το 2004, 11 Μαρτίου συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα το 5.000, το οποίο έχει να κάνει με 250 άτομα στην Λετωνία που τους αφαιρέθηκε το δικαίωμα της ηθαγένειας. Είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό σε σχέση με τον πληθυσμό στην Λετωνία. Σας υποβλήθηκαν πολλές κατηγγελίες για την περίπτωση αυτό. Πρόκειται για μια παρανομία που έγινε και το θέμα αυτό δεν έχει επιληθεί ακόμα. Δεν νομίζετε λοιπόν ότι είναι άδικο κύριε Διαμαντούρο Νομίζω ότι έχει ανοίξει το κουτί της Πανδώρας, κανείς όμως δεν μπόρεσε και δεν προσπάθησε ακόμα να επιλύσει αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Για δύο λεπτά ο κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που σας βλέπω και πάλι στο Προεδρείο. Ιδιαιτέρως χαίρομαι. Εύχομαι να είστε πάντα γερός και δυνατός. Κυρίες και κύριοι, την περίοδο αυτή, ιδιαίτερα στις χώρες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες λόγω της οικονομικής κρίσης, βλέπουμε την κρίση και στην εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε το σκεπτικισμό με τον οποίο πολλοί συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό άλλωστε η χρονιά αυτή που την έχουμε αφιερώσει στους πολίτες μας είναι το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών φέτος και έχει πρωταγωνιστήσει και αντιπρόεδρος τη Επιτροπής για να το έχουμε αυτό η κυρία Ρέντινγκ. Όλοι κουβεντιάζουμε, όλοι συζητάμε πώς μπορεί να ενισχυθεί η θέση και η σχέση των πολιτών ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή όλα αυτά τα χρόνια έχει παίξει καθοριστικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή. Σωστά στην εξαιρετική έκθεσή του ο εισηγητή μα, ο κύριο Αλαβράκο, αναφέρεται όχι μόνο στα πεπραγμένα του 2012, ιδιαίτερο σε αυτήν την έκθεση, αλλά και κάνει κατά κάποιο τρόπο μια αποτίμηση τη δεκαετία. Γιατί πράγματι τα χρόνια αυτά ο θεσμό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ενισχύθηκε. Εκείνο που προσωποποίησε αυτόν τον θεσμό ήταν ο κύριο Νικηφόρο Διαμαντούρο, ο οποίο κατά κοινή ομολογία έκανε εξαιρετική δουλειά και είναι καθήκον όλων μα να συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτόν τον θεσμό τα επόμενα χρόνια, να στηρίξουμε και την διάδοχό του, την κυρία Ορέιλι, προς την κατεύθυνση αυτή. Είμαι πεπισμένος ότι το επόμενο διάστημα οι πολίτες θα, θα βρεθούν πιο κοντά στην Ευρώπη. Είμαι πεπισμένος ότι αυτά που κερδίσαμε μέχρι σήμερα με τον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή θα τα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο. Η ταχύτητα στην ανταπόκριση στα αιτήματα, η αμεσότητα με το διαδίκτυο και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκαν κάθε ε, όλα αυτά τα χρόνια. Ε, καλή δύναμη κύριε διαμαντούρο πραγματικά τιμήσατε ε, τον θεσμό όλα αυτά τα δέκα χρόνια. επιτρέψτε μου όμως να πω και κάτι τελευταίο αυτά τα χρόνια τιμήσατε και την πατρίδα σας την ελλάδα. σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο. Εφόσον έχουν μιλήσει όλοι οι ομιλητές, φτάνουμε στην διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑΗ. Ο κύριος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον διαμεσολαβητή μας. Σας ευχαριστούμε για αυτά τα δέκα χρόνια. Νομίζω ότι η θέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι πολύ ιδιαίτερη και ευαίσθητη όμως. Αν συνοψίζαμε το έργο σας, θα έπρεπε να πούμε ότι ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικό. Πιστεύω ότι ο διαμεσολαβητής είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε εμά και τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι κάποιος ο οποίος ασχολείται με τα προβλήματα των πολιτών, αλλά προσπαθεί να επιβάλλει και τη διαφάνεια στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτό λοιπόν βοηθάει τους πολίτες να βρουν την έξοδο από το δέδαλο της Ευρωπαϊκής Γραφειοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ και ό,τι καλύτερο για το μέλλον, κύριε Διαμαντούρο. Ευχαριστώ τον συνάδελφο. Επόμενη ομιλήτρια για ένα λεπτό, η κυρία Σμόλκομα. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Διαμαντούρο για το έργο του που φρόντισε να ενισχυθεί η διαφάνεια στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Το έργο του Ευρωπαίου Διαμασουλευτή είναι πολύ σημαντικό και κάθε άλλο παρεύκολο. Πρέπει να πούμε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν διευκόλυναν το ρόλο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Το είδαμε αυτό τα τελευταία χρόνια με τις καταγγελίες που έχουν κατατεθεί και το έργο του Ευρωπαίου Δημοσιολογητή δεν έχει ολοκληρωθεί σε όλες τις περιπτώσεις. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειάστηκε να διπλασιάσει τις προσπάθειές του τα τελευταία χρόνια. Οι υψηλές προδιαγραφές, σεβασμός των δικαιωμάτων των πολιτών πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας, γνωρίζοντας ε, μάλιστα, πόσο μάλλον δηλαδή τώρα που πολύ σύντομα θα έχουμε ευρωεκλογέ και θα ζητήσουμε τη στήριξη των πολιτών και την εμπιστοσύνη των πολιτών σε μας. Σας ευχαριστώ πολύ που δημοσιεύσατε και τον κώδικα διοντολογίας που ελπίζω ότι θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την διαφάνεια και την χρηστή διαχείριση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο. Αυτοί ήταν οι ομιλητές που είχαν δηλώσει για την διαδικασία Catch the Eye. Οπότε ερχόμαστε και πάλι στην Επίτροπο Ρέντινγκ εκ μέρους της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, 24 χρόνια βρίσκομαι εδώ, 10 χρόνια ως Ευρωβουλευτής και 14 χρόνια ως Επίτροπος. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω ότι ποτέ στη ζωή μου δεν ξαναείδα κάτι τέτοιο. Δηλαδή από όλε τις πλευρές, από όλα τα έδρα. όλοι να συμφωνούν και να επικροτούν το έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και των συνεργατών του. Είναι εκπληκτικό, όπως εκπληκτικό ήταν και το έργο σας κύριε Διαμαντούρο. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω, μόνο να απαντήσω σε μία ερώτηση που μου απευθύνθηκε. Εννοείται ότι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα υπάρχει περιθώριο για περισσότερο χρηστή διοίκηση. Οπότε Καλοδεχόμαστε τις παρατηρήσεις του Ευρωπαίδιου Μεσολαβητή και προσπαθούμε τις παρατηρήσεις του να τις εφαρμόσουμε και στην πράξη. Λαμβάνουμε υπόψη μας τις προτάσεις του και συνεργαζόμαστε με πολύ θετικό πνεύμα μαζί του και το ίδιο θα κάνουμε και με την διάδοχό του. Όσον αφορά τώρα τους κανόνες χρηστής δίκησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει την ανάλυση του υπάρχοντος κοινοτικού δικαίου για να δει κατά πόσο καλύπτονται όλοι οι τομείς ή όχι. Όλοι οι τομείς δηλαδή που έχουν να κάνουν με τη χρηστή δίκηση. Και βάσει της ανάλυσης αυτής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίσει κατά πόσο πρέπει να υπάρξει κανονισμός που να βασίζεται στο άρθρο 298. Εάν ναι, θα το πράξουμε μόνο όμως εάν φανεί ότι υπάρχει τέτοια αναγκαιότητα και από την μελέτη φανεί ότι δεν καλύπτονται όλα. Συνεπώς η Ευρωπαϊκή Επιτροφή πρέπει να ξέρετε ότι έχει θετική προσέγγιση, θέλει να κάνει τη δουλειά της και συνεχίζει να την κάνει. Προκειμένου να υπάρχει πλήρης διαφάνεια παρόλα αυτά, πρέπει να σας εξηγήσω ότι μια τέτοια ρύθμιση δεν μπορεί να χρησιμεύσει για να θέσει κανόνες σε σχέση με άλλα άρθρα της συνθήκης πέρα του 298, για παράδειγμα πρόσβαση στα έγγραφα που υπάρχει κανονισμός ή δημοσιονομικοί κανονισμοί. Συνεπώς εδώ μιλάμε για τη χρηστή διοίκηση και μόνο. Τα άλλα προβλήματα πρέπει να λυθούν σε άλλο επίπεδο. Και βλέπω από τον ε, Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να γνέφει καταφατικά, άρα είναι σωστή η προσέγγιση αυτή. Συνεπώς, είναι πολύ καλό να έχουμε ένα ισχυρό θεσμό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Είναι θετικό για όλα τα θεσμικά όργανα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διαμεσολαβητά. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Επίτροπο. και ε, θα παρεκκλίνω λίγο από τον ε, ρόλο μου και θα θέλω κι εγώ να συνταχθώ με αυτή την διακομματική ας πούμε τάση για να συγχαρούμε όλοι μαζί τον κύριο ε, Διαμαντούρο για την εξαίρετη δουλειά που έχει κάνει θα τον ευχαριστήσω ε, και εγώ προσωπικά λοιπόν. Αυτό βέβαια που θα πρέπει να πω πάνω απ' όλα είναι ότι ήταν ένας εξαίρετος ε, διαμεσολαβητής για τους πολίτες. Ε, και με αυτά τα λόγια δίνω και πάλι το λόγο στον κύριο Διαμαντούρο. <clears throat> Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι συμμερίζομαι απόλυτα, μάλλον ότι, ναι, συμμερίζομαι τα σχόλια των συναδέρφων σχετικά με την επιστροφή σας εδώ. Χαίρομαι και εγώ πολύ που σας ξαναβλέπω εδώ. Επιτρέψτε μου τώρα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά την ουσία του θέματος που συζητάμε και να απαντήσω στις παρατηρήσεις σας σχετικά με το θεσμό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το γραφείο μου. Όσον αφορά την ουσία των σχολείων, τα εξή. Πρώτον, είμαι ευγνώμων στην κυρία Ρέντινγκ, η οποία ενημέρωσε το σώμα για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει πολύ σοβαρά τη δυνατότητα να υιοθετήσει αυτό το οποίο τελικά θα είναι το δίκαιο για την ε, διοικητική μεταρρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βασίζεται στο άρθρο 298. Είναι πολύ θετικά νέα αυτά. Η διαδοχός μου βέβαια είναι εκείνη η οποία θα συνεργαστεί μαζί σας, θα σας συμβουλεύσει για να προχωρήσετε σε αυτή τη διαδικασία. Κυρία Ρέντινγκ, το βασικό είναι οι πολίτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με σαφήνεια να καταλαβαίνουν πώς λειτουργούν τα πράγματα και όχι να μπερδεύονται ανάμεσα σε πολλά και διαφορετικά μέσα τα οποία προσπαθούν να πετύχουν τη χρηστή διαχείριση. Η απλοποίηση λοιπόν που προσπαθεί να πετύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάτι πολύ θετικό. Το ξέρετε κι εσείς από την εμπειρία σας ότι η σαφήνεια σημαίνει καλύτερα αποτελέσματα και πιστεύω ότι όντως θα προχωρήσετε προς αυτήν την κατεύθυνση και σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια που κάνατε και είπατε ότι θέλετε να ενισχύσετε και τις ρυθμίσεις για το περιβάλλον. Πράγματι και εγώ χαίρομαι για τις βελτιώσεις που έγιναν σε σχέση με το αεροδρόμιο της Βιέννης. Οπότε επαναλαμβάνω τις ευχαριστίες μου και ελπίζω και εγώ ότι η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τη διάδοχό μου για να προωθήσει νέα ε, νέες νομοθετικές διατάξεις οι οποίες θα ενισχύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στείλει το μήνυμα στους Ευρωπαίους πολίτες ότι κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και ότι τους βοηθάει. Τώρα επιτρέψτε μου να πω επίσης στον κύριο Μίνσκι. Κύριε Μίνσκι, μετά από εννέα χρόνια πρέπει να ομολογήσω ότι δεν θυμάμαι ακριβώς τι έγινε το 2004. Αυτό όμως που πρέπει να σας πω είναι ότι δεν θυμάμαι το γραφείο μου να πήρε καταγγελία για αυτό το θέμα σε εθνικό επίπεδο στην Λετωνία. Ότι έγινε μάλλον σε εμά η καταγγελία αυτή. Νομίζω ότι έγινε στη Λετωνία η καταγγελία αυτή. Αλλά το γραφείο μου είναι στη διάθεσή σας εφόσον θέλετε ευχαρίστως να το εξετάσω και το προσωπικό μου αλλά και η κυρία Ορέλη σίγουρα θα μπορέσει να σας απαντήσει πιο υπεύθυνα από αυτά που μπορώ να σας πω εγώ γιατί μετά από τόσα χρόνια ομολογώ ότι δεν θυμάμαι ακριβώς. Τέλος, πριν περάσω σε πιο γενικά σχόλια, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ματσόνη για την στήριξή της στο πρόσωπό μου και για την στήριξη που ολόκληρη η Επιτροπή Αναφορών μου προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι πραγματικά ευγνώμων. Τώρα κύριε Πρόεδρε. Είναι δύσκολο να πω οτιδήποτε άλλο από το ότι είμαι ειλικρινά ενθουσιασμένο από τα σχόλιά σας, από τη στήριξη που είχα όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζω να έχω από όλους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω με ευγνωμοσύνη και ταπεινοφροσύνη. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι όλα αυτά τα καλά σχόλια έχουν να κάνουν με το θεσμό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και έχουν να κάνουν επίσης και με την αύξηση των υποχρεώσεων που ανέλαβε και που πρέπει να αναλαμβάνει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής προσπαθώντας να προχωρήσει στο μέλλον και να βοηθήσει τους Ευρωπαίους πολίτες και να βοηθήσει και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να περάσουν σε μια πιο θετική νοοτροπία. Όλα αυτά, από εδώ και πέρα, τα αναλαμβάνει η κυρία Ορέλη. Και μετά τα λόγια που ακούστηκαν εδώ, ξέρει η κυρία Ορέλη τι έχει να αντιμετωπίσει, ότι έχει την εμπιστοσύνη σας, ότι έχει τη στήριξή σας. Πολύ σημαντικό αυτό. Κάποιοι από εσά είπαν ότι είναι ειδικό θεσμικό όργανο ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Εγώ εδώ θα ήθελα να σας θυμίσω κάτι το οποίο έκανε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και πώς βοήθησε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στην Τουρκία και συναντήθηκα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και υπουργούς επί τη ευκαιρία του θεσμού του Τούρκου διαμεσολαβητή που επιτέλους εγκαθιδρύθηκε και βοήθησα και εγώ σε αυτό πράγματι όλα αυτά τα χρόνια. Είπα λοιπόν και στον κύριο Ορτογκάν και στον κύριο Γκιούλ και στους υπουργούς ότι ο διαμεσολαβητής είναι πράγματι ένα πολύ ιδιαίτερο θεσμικό όργανο. Και γιατί? Γιατί έχει την υποχρέωση να λέει την αλήθεια στην εξουσία. Να λέει δηλαδή στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο τι ακριβώς συμβαίνει και πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να ξέρουν ότι ο διαμεσολαβητής τους θα τους λέει τα πράγματα όπως έχουν. Και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχει ο διάλογος. Και γι' αυτό και είμαι ευγνώμων σε εσά για το διάλογο αυτό που είχαμε μεταξύ μας όλα αυτά τα χρόνια. Τέλος. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα κάπως πιο λεπτό. Έχω έρθει σε επαφή με ειδικού γλωσσολόγους και τα λοιπά από τις σκανδιναβικές χώρες. Στη Σουηδία λοιπόν και στην Ισλανδία ο όρος Όμπουτσμαν δεν έχει ούτε ε, δεν έχει γένος, δεν είναι ούτε θηλυκό ούτε αρσενικό. Τώρα βέβαια έχουμε την Ευρωπαία διαμεσολαβητή. Δεν ξέρω πώς θα χειριστεί αυτό το θέμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς θα αποκαλεί την κυρία Ορέιλη. Πάντως σας λέω ότι έκανα κάποιες έρευνες και από εκεί και πέρα εσείς θα αποφασίσετε μαζί με την κυρία Ορέιλη ποιος θα είναι ο σωστός τίτλος, πώς θα πρέπει να απευθύνεστε σε αυτήν. Αλλά ελπίζω να αποφύγετε αυτό που έχει γίνει από την άλλη μεριά του Ατλαντικού που τώρα έχουν φτιάξει και ρήμα. Ε, από το Ombudsman. Η... Όπως και να έχει πάντως το πράγμα, να ξέρετε ότι είμαι ευγνώμων σε εσά για τη στήριξή σας και τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ και πραγματικά Φροντίστε την επαφή αυτή με την κυρία O'Reilly, Mrs. O'Reilly, λέει στα αγγλικά ο κύριος Διαμαντούρος, προκειμένου η καλή συνεργασία να συνεχιστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον ε, διαμεσολαβητή. Επόμενος ε, έχει το λόγο ο κύριος ε, Σαλαβράκος για δύο λεπτά ως εισηγητής. Να σας πω ότι για να σεβαστούμε την ημερήσια διάταξη ε, είχαμε μία ανοχή για τις υπερβάσεις χρόνου, όμως ε, στις επόμενες ομιλίες θα είμαι πολύ αυστηρός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εξέλιξη της συζητήσεως μου επιτρέπει να κάνω την σύνοψή της με μια ομοιρική λέξη. Ένεπε το Ευρωκοινοβούλιο, ένεπε στον απερχόμενο μεσολαβητή την πλήρη συμπαράστασή του και την πλήρη αναγνώριση του έργου του. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο θεσμός του μεσολαβητή είναι δικαιακός. Δεν είναι δικαστικός. Και επειδή είναι δικαιακός θεσμός είναι ακόμη πιο δύσκολος. Διότι δεν είναι αναγκαστές οι αποφάσεις του μεσολαβητή. Οι δικαστικές αποφάσεις εξαναγκάζονται εκτελούνται. Οι αποφάσεις του Μεσολαβητή αποδίδουν μια δικαιοσύνη η οποία γίνεται σεβαστή από το κύρος του προσώπου και από την αρθότητα των αποφάσεων. Και σε αυτά είχαμε επιτυχία την τελευταία δεκαετία. Οι Ευρωπαίοι πολίτες οι οποίοι είναι οι χρήστες αυτού του θεσμού εξητούν μια διαβίωση σε καλό κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο και πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία διαβίωση σωστή εάν δεν υπάρχει δικαιοσύνη. επομένως πρέπει με δικαιοσύνη να αντιμετωπίσουμε τους ευρωπαίους πολίτες. φοβάμαι ότι όταν γεννώνται προσχήματα ή δημιουργούνται προσχήματα για κυβερνητικές αυθαιρεσίες κάτι δεν πάει καλά και η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει πολλά προσχήματα για κυβερνητικές αυθαιρεσίες σε όλα τα επίπεδα κυβερνήσεων πιστεύω όχι μόνο στην ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. πρέπει να το προσέξουμε. η εξήτηση τη δικαιοσύνης από τους πολίτες της ευρώπης είναι πιο έντονη διότι σήμερα δυστυχώς στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται και ο ρόλος της κυρίας ε, επιτρόπου είναι σημαντικός. Κλείνοντα, δεν θέλω να μακρηγορήσω ευχαριστώ και για τη συμπαράσταση όλων των πολιτικών ομάδων προ την ε, έκθεσή μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι λοιπόν τελειώνει η συζήτηση για αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 12. Επόμενο σημείο στη ημερήσια διάταξη, η έκθεση του κυρίου Χέντελ για